Αγαπητοί συναδελφοί, θα ολοκληρώσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου και προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κλάς. Η κυρία Ρόιτ, το βαγιά, ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να προσδορίσουν ένα σχέδιο δράσεως και χρονοδιάγραμμα για την κατάρριξη χρήση των φυτοφαρμάκων και ζώνες ασφαλής για την προστασία των πόσιμων υδάτων. Πρόκειται για μια πρόταση αποδεκτή και πιστεύω πρόταση που θα τυχεί της υποστήριξης των Ευρωπαίων πολιτών και την υπερψήφιση. Η κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω ότι ψήφισα υπέρ αυτής της συμβαστικής πρότασης διότι θεωρώ ότι είναι λογικό να έχουμε μια ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που ισχύουν σε διάφορα κράτη-μέλη και ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν ε, την κατάρτιση και την εκπαίδευση με έναν πολύ καλό τρόπο έτσι ώστε έχουμε σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων. Άλλε χώρε όμω δεν το κάνουν αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι καλό θα είναι να έχουμε μια ε, νομοθεσία η οποία να, έχουν, ε, να, ναι, η οποία να εξασφαλίζει μια ορθολογική χρήση αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι γίνεται με του ψεκασμού κτλ. Τέλο πάντων θεωρώ ότι είναι μια καλή αντιμετώπιση και συγχαίρω την εισηγήτρια, η κυρία Ντόιλ.

Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ υποστήριξα την ε, έκθεση αυτή. Όντω, χρειαζόμαστε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα φυτοφάρμακα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί. Η έκθεση κλάσα περιορίζει την, ε, την άλογη χρήση των φυτοφαρμάκων. Όμω το πρόβλημα είναι και στην έκθεση, ε, υπάρχει και στην έκθεση Μπράγερ για την διάθεση φυτοβροσευτικών προϊόντων. Το πρόβλημα είναι όμω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μα και την αγορά στην έκθεση θα πρέπει ε, να δούμε και πόσο το να είναι ε, ένα προϊόν στην αγορά από μόνο του δεν αποτελεί κίνδυνο. Ε, ο κίνδυνος για τα φυτοφάρμακα υπάρχει εάν τυχόν δεν γίνεται σωστή χρήση, εάν ο δεν είναι αγνοείται και δεν χρησιμοποιείται σωστά, εάν δεν αποθηκεύονται σωστά τα φυτοφάρμακα. Επομένως, η ναι μεν είναι καλό να χρησιμοποιούνται λιγότερα φυτοφάρμακα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον αριθμό των ψεκασμών που γίνεται και με το διάλειμμα το οποίο χρησιμοποιείται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο, ε, στην επόμενη έκθεση για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η κυρία Ρόιτεβα. Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στα όσα υπόθηκαν εχθέ στην Ολομέλεια. Εγώ υποστηρίζω τη νέα νομοθεσία γιατί είναι ένα καλό μέσο και θα εξασφαλίσουμε πιο ασφαλεί τρόπους παραγωγής φαρμάκων και ακόμα ένα βήμα προόδου με την αμοιβαία αναγνώριση των ε, φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται αναγεωγραφική ζώνη. Επίσης, θετική εξέλιξη ήταν η κατάρτιση των καταλόγων με τις καρκινογενείς και λοιπές ε, νευροτοξικές ή άλλες ουσίες που ε, στηρίζεται στις επιστημονικές, στα επιστημονικά πορίσματα. Πρόκειται για ουσίες που μπορεί να έχουν χαμηλά ποσοστά. Σας υπενθυμίζω όμως ότι τα προϊόντα θα πρέπει να υπάγονται στις αντίστοιχες απαιτήσει ασφάλειας. Θα ήθελα επίσης να δώσω Στις άλλες ε, εκθέσεις για τις οποίες έχουν, έχει λήξει βέβαια η συζήτηση, αλλά θα σας δώσω γραπτές επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ κυρία Γουόλης, πρόεδρε. Θα πρέπει να κάνω μια, να σας ομολογήσω ότι από παιδί αντιπαθώ τον Αρακά και όμως προέρχομαι και εκπροσωπώ από τη, μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής Αρακά του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμφωνώ λοιπόν με την έκθεση, με τους στόχους της, με τους στόχους της νομοθεσίας που είναι η προαγωγή τόσο της υγείας του περιβάλλοντος, του καθαρού περιβάλλοντος αλλά και της υγείας, της δημόσιας υγείας, της υγείας των πολιτών. Αλλά φοβούμε ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μακροπρόθεσμα μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής, ιδιαίτερα από την περιοχή μας και γι' αυτό ε, δήλωσα την αποχή στην ψηφοφορία, ύστερα από πολύ ωρίμη σκέψη. Βλέπω ότι τα οι επιλογέ που έγιναν μέσα στην έκθεση ήταν εσφαλμένε τελικά, γιατί δόθηκαν τόσε πολλέ πληροφορίε, αντιφατικέ μάλιστα, που και, εμεί, και εγώ όπω και άλλοι θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία για μια τρίτη ανάγνωση, την συνδιαλλαγή δηλαδή, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε πρόσπιση κάθε συμφέρον κάθε πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ. Θεωρώ ότι είναι δύσκολη, σκληρή απόφαση που χρειάστηκε να λάβουμε. Ήταν βέβαια πολύ καλή και επικοδομητική η προετοιμασία της εκθέσεως και στόχος μας ε, η προστασία σε ύψιστο βαθμό της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Πλην όμως ε, τρέφω πολλές ανησυχίες ως προς την ε, ορθότητα των αποφάσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις για επικίνδυνες ουσίες. Τώρα στηριζόμαστε στο κατά πόσον μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο μία ουσία χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπόψη τον πιθανό, την πιθανή έκθεση στην ουσία αυτή. Χρειαζόμαστε στοιχεία επιστημονικά για να μπορέσουμε να λάβουμε τι αποφάσει. Και από τα στοιχεία που έχω εγώ, από τι συνομιλίε με πολίτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνω ότι ένα από τα θέματα που διαρκώ του απασχολούν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ομοθοσία τη έρχεται δυσανάλογα να παρέμβει στη ζωή του. Και μπορεί βέβαια να προσφέρει ευελιξία αυτή η έκθεση, αλλά θα θέλαμε περισσότερη ευελιξία. Και πάνω απ' όλα θα θέλαμε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία για να στηρίξουμε τι αποφάσει μα. Βεβαίω η αρχή τη πρόληψη θα πρέπει να υπερισχύει και δεν το λησμονώ αυτό, αλλά όποια αποφάση λαμβάνουμε να στηρίζεται πάνω σε επιστημονικέ αποδείξει και τεκμήρια που δεν είχαμε σε αρκετό βαθμό στο πεδίο αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ζούλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο χρήση των φυτομαρμάκων είναι μία ανάγκη. Η προστασία του περιβάλλοντο, η προστασία τη δημόσιας υγεία προχωρούν μαζί, αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών. Ε, ναι, μεν καλωσορίζω του στόχου ε, τη έκθεση Μπράγερ ότι θα πρέπει ε, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία δεν ε, συμφωνώ με ορισμένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται και η, η, η περιοχή από την οποία προέρχομαι, το Midlands, Midlands, έχουμε με φοβερές αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικά θα είναι, κάτι, θα είναι αυτά τα μέτρα και όντως πιστεύω ότι δεν έχει γίνει μια αξιολόγηση των συνεπειών από την Κομισιόν και τι σημαίνουν όλα αυτά για την γεωργία αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων σε όλο τον κόσμο. επομένως δεν χρειάζεται να εισάγουμε αυτή τη στιγμή εμείς μέτρα τα οποία θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα στην παραγωγή των τροφίμων. Γι' αυτό είχαμε πει ότι θα έπρεπε να γίνει και μια λεπτομερής και ενδελεχή εξέταση των, αξιο... των συνεπιών. Κυρία Μαγκίνες, Πρόεδρε, όπως και άλλοι συνάδελφοι θεωρώ ότι ήταν ε, το θέμα αυτό πάρα πολύ δύσκολο και η Wallis ανησυχούσε για, τα, για, τα, για, τα, για τον Αρακά. Σκεφτείτε εμείς τι γίνεται με τις πατάτες στην Ιρλανδία. Ε, πιστεύω ότι ε, το αρχικό πακέτο ήταν πολύ πιο δύσκολο και συγχαίρω όλους όσους ε, εργάστηκαν για να έχουμε το πακέτο αυτό που ψηφίσαμε σήμερα, ε, θα πρέπει οι γεωργοί και οι αγρότες να πιέσουν την χημική βιομηχανία έτσι ώστε να παράγουν πιο ασφαλή προϊόντα για να συνεχίσουν και οι αγρότες να παράγουν ε, τα τρόφιμα τα οποία χρειαζόμαστε. Όσον αφορά τις εισαγωγές των τροφίμων, η Κομισιόν θα πρέπει να ικανοποιήσει μια πάρα πολύ σωστή ανησυχία που έχουν οι αγρότες. Είναι ότι δηλαδή εμείς ε, δεν χρησιμοποιούμε σε επικίνδυνες ουσίες. Οι αγρότες όμως των τρίτων χωρών συνεχίζουν να τι να χρησιμοποιούν αυτές τις επικίνδυνες ουσίες. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Ο κύριος Μότ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατεψήφισα την έκθεση αυτή απλώς και μόνο γιατί η πρόταση ε, την, την, την, έκλεψαν, την έκλεψε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εδώ υπάρχει μία ένωση διαφορών, αν θέλετε, και ένας τομέας ε, όπου χρειάζεται ποικιλία και διαφορά, διαφορετικότητα είναι αυτός εδώ. Ήταν, είναι βασικά αυτό το θέμα γεωργικό και όμως ο Επίτροπος για την Γεωργία, ο Δανός Επίτροπος για την Γεωργία ήταν απόν σε όλες τις συζητήσεις. Και ποιο είναι, ποια, είναι ο λόγος, είναι γιατί υπάρχει μια σύγκρουση ε, συμφερόντων, διότι απαγορεύθηκε στην Δανία να παρεύουν στο νερό από τη στιγμή που αντλείται. Λοιπόν, ε, εδώ είναι σαν να θεωρούμε ότι οι γεωργοί δεν ξέρουν τι να κάνουν και πρέπει να τους πούμε τι θα κάνουν. Εδώ νομίζω ότι έχετε ε, προσφέρει ένα όπλο σε αυτούς που μισούν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ντόιλ. Νομίζω ότι ακούστηκαν διάφορες υπερβολές και διάφοροι φόβοι και ήταν δύσκολο να, να διακρίνουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι, ποια είναι η επιστημονική φαντασία. Ναι, μεν καταλαβαίνω ποιες, είναι οι ανησυχίε και για την παραγωγή των, για για της πατάτας, του αρακά κτλ. Καταλαβαίνω τα συμφέροντα και τις ανησυχίες βασικά των γεωργών εγώ θεωρώ ότι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ξαναρχίσει η διαδικασία συνένεσης, συμφιλίωσης για αυτό το, για αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει η χημική βιομηχανία να συνεχίσει τις προσπάθειες για να προσφέρει εναλλακτικά προϊόντα. Κύριος Καμάλ, ευχαριστώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και την διαλεκτική με τον ε, τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Ε, μιλάμε για δημοκρατία και αγνοούμε τις, ε, τα αποτελέσματα δημοψηφισμάτων. Μιλάμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους αγρότες σε φτωχές χώρες. Τώρα όμως, σαν αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, θα απαγορεύσουμε τις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από από γεωργούς που έχουν χρησιμοποιήσει τα φυτοφάρμακα τα οποία έχουν απαγορευτεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση ε, να σκεφτόμαστε και στο μέλλον τις ε, απροσδόκητε και τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των ε, ενεργειών μας. Πιστεύω ότι βιαστήκαμε, ότι χρειάζεται και μια τρίτη ανάγνωση και πρέπει να γίνει μια ενδελεχής επιστημονική αξιολόγηση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Ο κύριος Ήτον Χάρις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ προσπάθησα να υπονομεύσω τη συμβαστική λύση καταψηφίζοντας στην έκθεση, αλλά να σας διαβάσω μια επιστολή για να εξηγήσω. Πρόκειται για μια επιστολή ενός γεωργού από την περιοχή μου. Ανησυχώ ιδιαίτερα. Έχω χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτοπροστασία όλα αυτά τα 40 χρόνια που είμαι αργρότη. Ε, ανησυχώ και προστατεύω στον βαθμό του δυνατού και τη δική μου βέβαια υγεία, τη δημόσια υγεία, αλλά και των ζώων τη περιοχή και, και το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, το να απαγορεύεται η χρήση ορισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα των μικητοκτόνων, ε, με βάση όχι επιστημονική ω κριτήριο, ε, ανησυχώ ιδιαίτερα ότι δεν θα επιτρέψει να συνεχίσω την δουλειά μου ω γεωργό εδώ. Πρόκειται μια επιστολή η οποία μοιάζει πολύ με άλλε εκατοντάδες που έχω λάβει από αντίστοιχου γεωργού από την περιοχή, από το Λέστερ, από το Nottinghamshire, από διάφορε επαρχίε τη περιοχή μου και γι' αυτόν τον λόγο καταψήφισα την πρόταση. Η κυρία Σίνοτ, τελευταία ομιλητρία. Τώρα που τέλειωσε η ψηφοφορία και τώρα που ακούστηκαν τα επιχειρήματα, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα στοιχείο κοινό στη συζήτηση, τόσο εδώ όσο και στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Η δυσπιστία απέναντι στον αγρότη. Η εντύπωση που εξέφρασαν ορισμένοι ότι ο Γεωργός προσπαθεί να καταστρέψει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία. Αυτό αντιβαίνει σε ό,τι γνωρίζω εγώ για, την, για τον ρόλο του Γεωργού, ο οποίος εκατοντάδες χρόνια, τουλάχιστον στην Ιρλανδία, αγωνίζεται, διατηρεί και προστατεύει το περιβάλλον, το διατηρεί καθαρό. Αποτελεί την πηγή της υγείας γιατί παράγει καλά προϊόντα, φαγητό καθαρό, πάνω στο οποίο στηρίζουμε και εμείς τη δική μας υγεία. Και θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τον Γεωργό παντού, ο οποίος με όλες τις σκληρές συνθήκες, το, τις ε, κλιματολογικές, ε, την ε, απαγόρευση των φυτοφαρμάκων και βέβαια την, γεωργική, την ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Συνεχίζουμε στις 3 με, τις, ε, με την έκθεση για τα βιομετρικά στα διαβατήρια. Διακόπτουμε τώρα τη συνεδρίαση.